Δίνω τον λόγο στον κύριο Αλέν Καντέκ, τον εισηγητή, για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, επί δύο μήνες διαπραγματευτήκαμε τα μέτρα που θα πρέπει να ε, εισαχθούν για να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, το οποίο ανατρέπει, θα έλεγα, τους κανόνες της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Ανέκαθεν σημειώνα και σημειώνω και σήμερα ότι θα είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί το μέτρο της εκφόρτωση κυρίως για τα πολύ εξειδικευμένα αλλιεύματα και για την ερασιτεχνικού τύπου αλλία. Σας εκλυπαρώ κύριε Επίτροπε, όταν ε, οι υπηρεσίες σας προβαίνουν σε σχεδιασμό νομοθετικών μέτρων θα πρέπει να υπολογίσουν και τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειές τους. Το να υποχρεωθούν οι αλείς να εκφορτώνουν κάθε αλίευμα σε κάθε έξοδο ε, μπορεί να έχει κάποια λογική, δηλαδή ενθαρρύνεται ο επαγγελματία τη Ελία να γίνεται πιο επιλεκτικό. Έστω. Στην πράξη όμω είναι πολύ δύσκολο, όπω σα έλεγα τώρα. Και το μας μέλημα λοιπόν είναι προφανώς να του τους αλληλευτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και μια αλληλευτική δραστηριότητα βιώσιμη και εξασφαλίζοντας επιλεκτικότητα των ε, συστημάτων της αλίας. Έχουμε μπορέσει χάρη στην έκθεσή μας να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες της προτάσεως. Καταρχάς θα πρέπει κάθε χρόνο να ε, καταγράφονται σε μια έκθεση που θα δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι συνέπειε για του αλληλεί. Αυτό χάρη στα προγράμματα, στα στοιχεία που θα διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη και από την 1η Ιανουαρίου μόνο του 2017 θα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό. Άρα θα έχουν δύο χρόνια, ενάμιση περίπου χρόνο για να προσαρμοστούν οι αλληλεί. Οι δε προτάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται από του οργανώσει των παραγωγών. Διευκόλυνση τη. Ε, αποθήκευσης και της εκφόρτωσης του γόνου ε, θα πρέπει να οργανωθούν, θα πρέπει να υπάρχει πιο ελαστική διάταξη νομοθεσία σε σχέση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποθήκευση επί του σκάφους και δεν θα υπάρχει δορυφορική τηλεεπιτήρηση στην τελευταία μα συζήτηση είχατε μιλήσει, στην προηγούμενη συζήτηση έγινε λόγο για το πολιετές πρόγραμμα για τη Βαλτική. Πολύ σημαντικό, όπω υπόθηκε, γιατί είναι το πρώτο το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο τη κοινή ελευτικής Πολιτική για την Αλία, που όπω είπε και ο κύριο Αλφρόντε και εσεί όμω, κύριε Βέλα, θα αποτελέσει ένα υπόδειγμα για τα λοιπά σχέδια αλίας και ε, διαχείριση Αλία. Ωστόσο, εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερο σχέση με το σχέδιο αυτό η στάση ορισμένων κρατών μελών τα οποία στο Συμβούλιο προσπαθούν να ε, καταστρατηγήσουν τις προνομίες του Κοινοβουλίου παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση της Βενεζουέλας που δικαίωσε το Κοινοβούλιο. Τα κράτη αυτά εξακολουθούν να αμφισβητούν τη διαδικασία της συναπόφασης για τα πολιετή σχέδια. Κοινή δήλωση της Γαλλίας και της Ισπανίας υπογραμμίζει και παραθέτω την ακαταλληλότητα της τακτικής Τη συνήθου νομοθετική διαδικασία. Και τα ίδια αυτά κράτη λένε ότι τα συμπεράσματα τη ομάδα κρούσεως για τα πολιετή ε, προγράμματα δεν έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο. Τι είναι αυτά και δεν έχουν διοργανικό καθεστώ. Τα συμπεράσματα ωστόσο έχουν ωραιότατα καθεστώ αμοιβαία εμπιστοσύνη σε σχέση με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Μια άσχεση εμπιστοσύνη όμω που η Ισπανία και η Γαλλία θέλουν να ανατρέψουν. Ω πρόεδρο τη Επιτροπή αλίας, καταδικάζω απερίφραστα αυτή την προσπάθεια παραβίαση των συνθήκων και καλό το Συμβουλίο που λυπούμε δεν είναι παρόν, εν τη σοφία του, να υιοθετήσει μια λογική θέση. Και δεν θα διστάσω να φτάσω στα άκρα για να υπερασπιστώ τι προνομίε του Κοινοβουλίου, εφόσον το Συμβούλιο θεωρήσει ότι προτιμάει να μετατρέψει την υπόθεση αυτή σε μια διοργανική αντιπαράθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπο Βέλα έχει το λόγο και τον καλό να περιοριστεί στα τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Αγαπητά μέλη, κύριε Καντέκ, όπως ξέρετε, ε, αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο για την πολιτική μας αυτή, ιδιαίτερα ως προς τις απορρίψεις που δημιουργούν ε, μία αρνητική εικόνα για την βιομηχανία και πλήττει διάφορα οικοσυστήματα, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα της αλίευσης. Η πρότασή σας που συζητάτε σήμερα και θα ψηφίσετε τη Δευτέρα αποτελεί ένα βασικό θέμα και θα δημιουργήσει ίσους όρους πρόσβασης ως προς τις ε, υποχρεώσεις φόρτωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αλέν Κατέκ και τους Σκιώδης για την ε, πολύ ε, καλή και σκληρή σας εργασία για να φτάσετε σε συμβιβασμούς. Και φτάσαμε σε μια συμφωνία που γίνεται αποδεκτή από όλους. Το κείμενο συμβιβασμού δέχεται βασικά στοιχεία της αρχικής μας πρότασης για να υπάρχει νομική σαφήνεια και για να μην υπάρχουν ασυνέπειες ως προς τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης και για να γίνει η σωστή εφαρμογή των κανόνων εκφόρτωσης. Η επόμενη φάση αφορά την Αλία στη Βόρεια Θάλασσα, στα ε, βορειοδυτικά και νότιο-ανατολικά ύδατα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε νομική, τη νομική ασφάλεια η οποία ε, αποτελεί πρόκριμα για αυτά τα σχέδια. Πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε και τις απορρίψεις και έχουμε μάθει και με τα πελαγικά, από τα πελαγικά είδη ως προς τις απορρίψεις και τις εκφορτώσεις. Οι εργασίες έχουν εντατικοποιηθεί και τώρα οι ομάδες των κρατών προβάλλουν κοινέ συστάσεις. Χρειάζεται διάδραση μεταξύ κομισιών και κρατών μελών. Κάτι το οποίο βαίνει καλός και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο πριν από την αρχή του επόμενου έτους. Τι γίνεται ως προς την εφαρμογή. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και τα κράτη-μέλη, βοηθώντας με μέσα που διαθέτουμε στην εργαλειοθήκη μας. Επίσης, είμαστε σε επαφή με το, τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πελαγικών Ιδών, έτσι ώστε να εποπτεύσουμε τις υποχρεώσεις εκφόρτησης Ακόμα και εάν δεν υπάρχει, δεν τίθεται σε εφαρμογή υποχρέωση όμνιμπους, ε, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αιτήματα διασάφης από κράτη-μέλη και πιστεύουμε ότι τα ζητήματα αυτά ήταν ίσονος σημασίας. Η συνεργασία είναι πολύ καλή μεταξύ επιθεωρητών των κρατών μελών και περιφερειακά και από τις πληροφορίες μας βλέπουμε ότι οι αλληλείς συμμορφώνονται με το γράμμα του νόμου. Εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτή την υπευθυνότητα που δείχνουν τα κράτη-μέλη και η βιομηχανία μέχρι τούδε και ελπίζουμε να ισχύσει κάτι τέτοιο και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και τώρα είμαστε στους ομιλητές και τις ομιλήτρες εκ μέρους των ομάδων. Πρώτα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού ο Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ανοίγουμε ένα νέο στάδιο στην Ευρώπη και θα πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε. Η εκφόρτωση όλων των αλλιευμάτων είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Σε μας αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Είναι η πραγματικότητα όμως και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε βιώσιμη αλία και για να το πετύχουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε πως θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα που θα κάνουν πιο εύκολα, ε, πιο εύκολη την εφαρμογή των μέτρων που έχουμε προτείνει. Οι αλληλείς να προσαρμοστούν καλύτερα στις νέες συνθήκες. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ καλό βήμα αυτό που πετύχαμε εν ώψη ε, των κυρώσεων που θα επιβάλλονται. Ε, νομίζω λοιπόν πως και οι αιτήσει μελέτες για το πώς λειτουργεί το μέτρο είναι θαυμάσιο. Καλή συμφωνία καλή συμφωνία ε, σε αυτό το πολύ κείμενο για τα όσα θέλουμε να πετύχουμε. Για την κοινή ελευθερική πολιτική, να σας πω πως ξεκινάμε τώρα, ο δρόμος μπροστά, μπροστά μακρύς. Μέτρα λοιπόν στα οποία θα συστρατευτούμε όλοι. Η υποχρέωση εκφόρτωσης, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το νομικό ε, μεταβατικό πλαίσιο που χρειαζόμαστε. Στα πλαίσια της αναθεώρησης μπορούμε να επιβάλλουμε και κάποιες τεχνικές ε, αλλαγές, για παράδειγμα τα τεχνικά περιφερειακά σχέδια. Αυτό το οποίο επήγει τώρα είναι οι επιχειρηματίες, οι πολιτικοί, οι αλληλείς, οι επιστήμονες και όλοι οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι φορείς να συζητήσουν πώς η υποχρέωση αυτή θα εφαρμοστεί στην πράξη γιατί περιμένουν με μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση, με πια ομοιογενή νομοθεσία, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα από τους πρώτους μήνες εφαρμογής. Σίγουρα έχετε καλή θέληση, το πιστεύω. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη διαδικασία αυτή έχουμε καλή θέληση, έτσι ώστε η ρύθμιση αυτή να είναι καλή για το χώρο της αλίας και να εξασφαλίζει το μέλλον αυτής της δραστηριότητας που είναι κομβική για την απασχόληση και το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια εκ μέρου των Σοσιαλιστών Δημοκρατών, κυρία Ουλρίκε Ρόντο, ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, οι υποχρεώσει εκφόρτωση εισήχθησαν για να απαγορευθεί η απόρριψη των ανεπιθύμητων αλλιευμάτων, που είναι ίσως πολύ μικρά ή όχι του ζητούμενου είδους. Αποτελούν όμως μεγάλη σπατάλη και κίνδυνο για την βιολογική πολυμορφία. Μεγάλες είναι οι ποσότητες των ε, παρεμπιπτών των αλλιευμάτων που απορρίπτονται στη θάλασσα. Πρέπει λοιπόν αυτό να αλλάξει. Και έτσι ε, πρέπει να έχουμε και τις διατάξεις για, τις ελάχιστες, για τα ελάχιστα μεγέθη και τις ε, διατάξεις για την απόρριψη και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο εισάγεται ώστε να ε, εφαρμόζεται απευθείας από τους αλληλείς, το ταχύτερο δηλαδή δυνατό, πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, η κυρία Τόμασιτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο κανονισμός Omnibus θα πρέπει να ισχύσει τώρα και να εναρμονιστεί με την υποχρέωση εκφόρτωσης για να μην υπάρχει μεγαλύτερο άχθος για τους αλείς. Θεωρώ ότι η επόμενη μεταβατική περίοδος που είναι διετή είναι σκόπιμη έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν οι αλείς. Βεβαίως ε, εγκρίθηκε εξαίρεση για την Κροατία ως προς την υποχρέωση εκφόρτωσης, ιδιαίτερα για το γάδο, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα δίχτυα δεν επιτρέπουν πολλές φορές από το να φτάσουμε σε απορρίψεις των παρεμπιπτόντων αλλιευμάτων. Αυτά τα προβλήματα όμως έχουν λυθεί εν μέρη και πιστεύω ότι φτάνουμε σε μια βιώσιμη πρόταση και θα την υπερψηφίσω. Σας ευχαριστώ. Ομάδα των Φιλελευθέρων. Κυρία Νίκολα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Φυσικά ο στόχος της υποχρέωσης εκφόρτωσης είναι ένας γενναιόδωρος ε, στόχος. Θέλουμε να μειωθεί η θνησιμότητα και να έχουμε μία προστιθέμενη αξία και να αποφύγουμε τις απορρίψεις. Δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε κατά τα τέλη του 2013 είχε μία μεταβατική περίοδο δύο ετών, άρα έχουμε καθυστερήσει. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες της ε, ΚΑΠ. Πιστεύω ότι είναι μια βιώσιμη πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά διότι οι υποχρεώσεις εκφόρτωσης αφορούν και την ίδια την επιτυχία της αλληλευτικής πολιτικής. Το Κοινοβούλιο είχε επικοδομητική στάση, προσπάθησε να απαλύνει αρνητικές συνέπειες και ελπίζουμε αυτός ο κανονισμός να στεφθεί από επιτυχία, αν και έχουμε πολλές αμφιβολίες, γιατί όπως είπε και ο ελεν κατεκ Κατέκ, δυστυχώς υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν είναι ευτυχή με αυτή την ε, προσέγγιση. Όμως εμείς θα πρέπει να την υποστηρίξουμε ε, για την ε, καλή, για το ίσιο πέρα της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια εκ μέλου τη ομάδα τη Γκουέντζιέλ, η κυρία Νί Ριάντα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κανονισμός αυτός παρουσιάστηκε για ποιο λόγο. Γιατί έχουμε συνέχεια απορρίψεις στη θάλασσα. Και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει περιβαλλοντική βιωσιμότητα και επίγει η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Γι' αυτό δεχόμαστε πως θα πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να ε, προστατεύσουμε και τους μικροαλληλείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν τους πολύ αυστηρούς κανόνες του κλάδου τους. Θέλω να είμαι σίγουρη πως ο κανονισμός αυτός δεν θα τους επηρεάσει αρνητικά. Είναι πολύ τεχνικός κανονισμός και για το λόγο αυτό πρότεινα τροπολογίες οι οποίες θα εξασφαλίσουν πως το διοικητικό βάρος αυτού του κανονισμού δεν θα βαρύνει υπερβολικά τους ε, μικροαλληλείς μας. Και προτείνω αυτή την υποχρέωση εκφόρτωσης να την υλοποιήσουμε σταδιακά. Θα πρέπει οι να βρεθούν στην καρδιά του κανονισμού γιατί πολύ συχνά αυτό δεν συμβαίνει. Και πολύ συχνά δεν ξέρουμε καν τι θα ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι εμείς εδώ να νομοθετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Έγκστρομ, εκ των Πρασίνων δεν είναι παρούσα και ως εκ του δίνω το λόγο για την ομάδα των EFTD, την κυρία Λουίς Μπόχς, μισή λεπτό. Ε, thank Ευχαριστώ πολύ. Η κοινή πολιτική αλίας είναι κακή πολιτική. Δεν είναι πρακτική, δεν είναι βιώσιμη, δεν δικαιολογείται. Στο τελευταίο, στην προηγούμενη θητεία προσπάθησαν να κάνουν μια μεταρρύθμιση και τελικά τι έκαναν, λιγότερο καταστροφική καταστροφή, δηλαδή σαν να άλλαξαν σειρά στις ξαπλώστρες του Τιτανικού. Δηλαδή, ναι, να σταματήσουμε τις απορρίψεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί αποτελεί ένα από τα χειρότερα σημεία ενός κακού συστήματος. Αλλά μια υποχρέωση εκφόρτωση που είναι μερική και περιορισμένη, δεν λύνει το πρόβλημα αυτό. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μην έχουμε πλέον αυτή την αυτούς τους τεράστιους ε, στόλους της Ισπανίας, της Γαλλίας που ε, ψαλπάρουν και ψαρεύουν στις θάλασσάς μας και μέχρι ε, να του σταματήσουμε θα πρέπει να πούμε στο Βρετανικό λαό πως οι Βρετανικοί πολιτικοί ηγέτες τους τους προδίδουν για μια φορά ακόμα γιατί οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Απλώς κάνουν μικροαλλαγές στο σύστημα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουντάν τώρα. Μία εγγεγραμμένη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η υποχρέωση εκφόρτωσης είναι μη εφαρμόσιμη. Δεν θα επιτρέπει δηλαδή να ε, κάνουν τη δουλειά του σωστά, κυρίως οι μικροί ερασιτέχνες ε, αλείς ε, θα επιβαρύνονται με επιπλέον χρόνο, κόστος σε καύσιμα για παραπάνω διαδρομές και επιπλέον τι σημαίνει εκφόρτωση, θα πρέπει να καταστρέφεται αυτό το με τον αλίευμα, θα πρέπει να ανακυκλώνεται, ποιο θα αναλάβει και ποιο επιπλέον θα αναλάβει το κόστο τη εκφόρτωση στην πραγματικότητα. Μια λογική λύση δεν ήταν να περιοριστούν τα απορρί... οι απορρίψει περιορίζοντας την παρεπίπτουσα αλία με νέες μορφές εξοπλισμού, με νέους τύπους εξοπλισμού. Πρέπει η αεραστεχνική αλία να εξασφαλίσει οπωσδήποτε παρεκκλήσεις και, ή και μία μεταβατική περίοδο για να προσαρμοστεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία θα επέτρεπε στον αεραστέχνη αλία να ενσωματώσει νέο εξοπλισμό προκειμένου να προσαρμοστεί στις κανονιστικές ρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά Κύριος Μιαρμόν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αυτή η πρόταση για τις απορρίψεις κάνει μια μεγάλη στροφή και είναι σημαντική. Οι αλληλείς θα πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια, το είπαμε, για να προσαρμοστούν τεχνικά σε αυτή την καινούργια διάταξη. Και στην περίπτωση της αλίας μικρής κλίμακας αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αύριο θα ψηφίσουμε ένα κείμενο όπου θα επιβάλλουμε μία νέα απαγόρευση των απορρίψεων και νέα εργαλεία. Εμείς πετύχαμε μία συμφωνία που αυτή τη στιγμή δίνει ένα περιθώριο ευελιξίας αλλά παρόλα αυτά επιβάλλει κάτι πολύ περιοριστικό υποχρεωτική εκφόρτωση όλων των αλευμάτων. Νομίζω λοιπόν πως εμείς Κάναμε προσπάθεια στην αρχική πρόταση Κομισιόν να τοποθετήσουμε κάποιες απαραίτητες αλλαγές έτσι ώστε ο Ευρωπαϊκός Στόλος να μπορεί αυτή την νέα υποχρέωση να την εφαρμόσει. Ο κλάδος αλληλείας χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Ξέρετε τι συμβαίνει στη Γαλλικία από όπου εγώ προέρχομαι που είναι η πρώτη, η μεγαλύτερη αλληλής της Ευρώπης. Εκφόρτωση όλων ε, των αλλιευμάτων σημαίνει άλλα εργαλεία, άλλα σκάφη. Και για την μικρή κλίμακα αλλιεία μπορεί να είναι ε, υπερβολικές οι δυσκολίες και αξεπέραστες. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της νέας απέτησης. Και θα ήθελα τέλος να σας πω πως η απαγόρευση των απορρίψεων θα φέρει κάποιες ε, ανισορροπίε στην αγορά στην Ευρώπη. Δηλαδή για τις ποσοστώσεις μεταξύ κρατών μελών. Πώς θα μοιράζονται. Μα είχαν βασιστεί σε ένα σύστημα το οποίο επέτρεπε τις απορρίψεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς να παραγγείλουμε μια μελέτη για να δούμε πώς θα κατανείμουμε τις αλληλευτικές ευκαιρίες από εδώ και στο εξή. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κυρία Κλάρα. Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτός ο κανονισμός Omnibus ε, που ε, επιβάλλει υποχρώσεις εκφόρτωσης θα πρέπει να ε, αναγνωρίσουμε ότι είναι ένας από τους πυλώνες της νέας ΚΑΠ. Πρέπει να τελειώσουμε με, το, με τις απορρίψεις και η νέα αλληλευτική πολιτική το κάνει. Υπάρχει λοιπόν η υποχρέωση για τη Βαλτική θάλασσα και τα πελαγικά είδη που θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Πρώτου. Πρόκειται για μία ε, ρυθμιστική αλλαγή που είναι ύψης της σημασίας, κάτι το καινοτόμο όπως είπαν και άλλοι. Θα πρέπει να σας πω κάτι κύριε Επίτροπε, ανησυχώ ιδιαίτερα γιατί ο ελευτικός τομέας έχει απειροελάχιστες πληροφορίες. Βεβαίως υπάρχουν λόμπι στις Βρυξέλλες, αλλά δυστυχώς οι αλευτικοί φορείς δεν έχουν πληροφορίες. Κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό και στο οποίο θα πρέπει να αρκεστούν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Τζέιμς Νίκολσον, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο αλληλευτικός κλάδος αντιμετωπίζει μεγάλες ε, προκλήσεις αντίστοιχε με τους άλλους τομείς, όπως η παράδειγμα, της γεωργίας και των τροφίμων. Ε, η πρόκληση είναι να κάνουμε περισσότερα για λιγότερο, λιγότερα έσοδα και πρέπει να εξασφαλίσουμε βιώσιμη και ευημερούσα ε, αλληλεία. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και τα πάντα η Ευρώπη, όπω και άλλοι ομιλητέ. Επίση, σήμερα η μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτική πολιτική στο Κέντρο του 2013 εισήγαγε μια υποχρέωση για του αλληλεί να εκφορτώνουν τα ε, παρεμπίπτοντα ε, αλλιεύματα με συνέπεια τελικά την απόρριψη των ε, ανεπιθύμητων αλλιευμάτων. Μακρυπρόθεσμα λοιπόν, οι προοπτικές για τον κλάδο της Αλίας θα είναι θετικές. Και χαίρομαι γιατί μπορεί το Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει περισσότερη ευελιξία σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στην μεταβατική περίοδο γιατί χρειάζεται δυνατότητα προσαρμογής στο μέλλον και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχηθώ ούριο άνεμο και ε, καλή επιτυχία, καλή δουλειά για τους αλληλείς της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιεν Χάτκτον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μην ξεχνάμε ότι η ΚΑΠ έχασε την αξιοπιστία της και ε, ακριβώς επειδή δεν είχαμε αντιμετωπίσει τις απορρίψεις στο παρελθόν. Θέλουμε να σταματήσουν οι απορρίψεις. Οι ίδιοι οι αλληλείς το επιθυμούν. Δεν θέλουν να ρίχνουν νεκρά ψάρια στη θάλασσα επειδή το επιβάλλει ο κανονισμός. Θεωρώ ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης θα πρέπει να ισχύσει μέσα στα πλαίσια μιας διαδικασίας περιφερειοποίησης. Δεν είναι τέλεια βέβαια όλα και θα είναι δύσκολο στα αμύκτα ήδη να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα στην Σκοτία. Χαίρομαι λοιπόν γιατί μας δίνεται χρόνο να ε, μπορέσουμε να προσαρμοστούμε, αλλά θα πρέπει να μειώσουμε τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα έτσι κι αλλιώς, έτσι ώστε η βιομηχανία να μην παραλύσει από αυτά τα, τα είδη τα οποία απορρίπτουμε. Και αυτό που έχει σημασία είναι να μειώσουμε την θνητότητα, όχι να μεταφέρουμε το πρόβλημα στη στερεά. Ευχαριστώ κύριε Μάρκο Αφρόντα, ένα λεπτό. Η υποχρέωση εκφόρτωσης έχει μεγάλη σημασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, απομακρύνουμε όλες τις απορρίψεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε μετά από ζωηρές συζητήσεις. Όμως το αποτέλεσμα είναι κατώτερο των προσδοκιών και στην ουσία μετουσίασε το ίδιο το κείμενο και τα αποτελέσματά του βασιζόμαστε και θα πρέπει να βασιζόμαστε σε επιστημονικά πλήρη στοιχεία. Γι' αυτό δεν έχει νόημα η εξαίρεση που μπήκε στον κανονισμό που ε, δεν επιτρέπει στη μικρή αλία τη στιγμή που τα είδη είναι κάτω των 50 κιλών. Πιστεύω λοιπόν ότι οι παραδοσιακοί αλίες ίσως να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν θα έπρεπε να έχουμε την ε, μεταβατική περίοδο των δύο ετών, αλλά με ε, ειδικέ ε, μνήε. Ευχαριστώ κύριο Σάντο για ένα λεπτό επίση. Νομίζω ότι αυτό ο κανονισμό πραγματικά θα ορίσει μια νέα αλλιευτική πολιτική η οποία θα σχετίζεται με μια ολιστική βιωσιμότητα θα λάβουμε υπόψη την αντιμετώπιση των απορρίψεων, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία ε, ιστορικά και πολιτικά. Η νέα αυτή όμως προσέγγιση θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τις μηδενικές ποσοστώσεις ιδιαίτερα στην ε, περίπτωση ορισμένων ειδών που θα μπλοκάρουμε γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη που υπάρχουν μηδενικές ποσοστώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ομιλητρία για τη διαδικασία Καριστία είναι η κυρία... πριν από το Καριστία είναι η κυρία Γκέρλινγκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερω που βρίσκομαι επιτέλου ε, σε θέση να υποστηρίξω την εκθέση. Ευχαριστώ τον κύριο Καντέ και την πολύ σκληρή δουλειά του. Ξέρω ότι ήταν δύσκολη. Ιδιαίτερα χαίρομαι, ε, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για τι καθυστερήσει τη υποβολή τη προτάσεω. Θα ήταν καλό να είχαμε εγκαίρω τον ε, κανονισμό, δηλαδή από την έναρξη του έτου για την απαγόρευση. Δεν έχουμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις προς τον κανονισμό όμνιμπους, προς τον πολυκανονισμό αυτόν δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι έχουμε πολύ, σημαντικά, πολύ σημαντικές απορρίψεις λόγω των καθυστερήσεων. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσει η Επιτροπή, να καταθέσει όλα τα τεχνικά μέτρα διατήρησης των αποθεμάτων, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, γιατί τώρα πια έχουμε λύσεις στα χέρια μας. Η μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής από το προηγούμενο κοινοβούλιο είχε ε, ως ένα από τα κύρια της επιτεύγματα την απαγόρευση των παρεμπιπτών των αλλιευμάτων και της απόρριψής τους, κάτι το οποίο ιδιαίτερα ε, κίνησε τον ενδιαφέρον των πολιτών, γιατί ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι ερχόνταν σε επαφή μαζί μου για να μου πούνε ότι ε, πρέπει να προχωρήσει αυτό το θέμα. Ας μην το ξεχάσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε τη δικασία Καρστιάη με πρώτο μιλητή, τον κύριο Βαλένσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. πρέπει κάποιος να βρούμε έναν τρόπο να εξαλείψουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι το 23% των εκφορτώσεων που επιτρεπόταν πριν ε, ε, πλέον έχει αλλάξει και όλοι οι αλλιέοι ε, πρέπει πλέον να εκφορτώνουν οτιδήποτε έχει εμπορική αξία. Υπάρχουν ε, αλλιεύματα τα οποία αλλιεύονται χωρίς ποσοστώσεις ή κάτω από το ελάχιστο μέγεθος. Αυτό φυσικά λοιπόν θα έχει πολύ καλές συνέπειες, θα μπορούσαμε να έχουμε αποτελεσματική χρήση των πόρων μας και θα ε, μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτή την ε, κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, έχετε την πλήρη υποστήριξή μου. Επόμενος ομιλητός, Uh, uh, Ο κύριος Πονσούλητσα για ένα λεπτό. Ε, πρόκειται για λάθος μάλλον. Εγώ δεν ζήτησα το λόγο στο ΚΑΤΣΔΙ για την υποχρέωση εκφόρτωσης. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος Ρίτσαρτ Κόρμπετ που ζήτησε το λόγο για αυτή τη ε, διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ ή όχι. Εντάξει. Ε, να σας παραλείψουμε και εσάς λοιπόν. Ο κύριος Νότης Μαριάς η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή στην αλλιευτική δραστηριότητα και το 2015 θα είναι έτος δοκιμής για την εφαρμογή της. Η πολιτική αυτή στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς θέτει τέλος στις απορρίψεις αλλιευμάτων στη θάλασσα. Όμως ο στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη αλλιευτικών αποθεμάτων πρέπει να στηρίζει ταυτόχρονα τη βιώσιμη αλλιευτική δραστηριότητα οφείλει να λάβει υπόψη της τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του κανονισμού στους μικροαλληλείς των κρατών μελών γιατί αυξάνει το κόστος λειτουργίας της μικρής κλίμακας αλληλείας και των παραδοσιακών αλλιέων. απαιτεί επιπλέον επενδύσεις και αύξηση του εργατικού κόστους. για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει μια σημαντική χρονική περίοδος προσαρμογής και πρόβλεψη χρηματοδοτικών ενισχύσεων και εργαλείων για την προσαρμογή των μικροαλλιέων στο νέο σύστημα γιατί το νέο πλαίσιο απαιτεί πέραν των άλλων και επενδύσεις για την αποθήκευση και επί του σκάφους. Ευχαριστώ. έχει το λόγο. εδώ πριν. Ε, αλλάξετε θέση με τον κύριο Σάντο. Είναι η σειρά σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη κύριε Επίτροπε. Ε, Μόλι έρχομαι από ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό, ε, το, ε, αυτό το κείμενο είναι τμήμα της μεταρρύθμισης της κοινή ελευθερικής πολιτικής και μιας προσπάθειας να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Και δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι αυτή της μηδενικής απόρρευσης, αλλά αυτή της υποχρεώση εκφόρτωσης. Ε, δεν αντιμετωπίσαμε το θέμα καταλήλω και λυπάμαι που δεν ε, αξιοποιήσαμε το χρόνο μας ώστε να ε, δώσουμε τις κατάλληλε λύσεις όσον αφορά την επιλογή των αλληλευτικών εργαλείων ώστε να μειώσουμε τη θνησιμότητα των αλληλευμάτων. Είναι κρίμα διότι επιλέγουμε και πάλι το δρόμο των αένων κυρώσεων. Ε, δυστυχώς η πλειοψηφία, όχι η δική μου, ε, ακολούθησε αυτή την άγουσα και δυστυχώς δεν βοηθάμε την κοινή αλληλευτική πολιτική με αυτά. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να τηρήσουμε αυτή την υποχρέωση, αυτή την απέτηση και δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει τη ζωή των ε, αλλιέων και την καθημερινή τους εργασία. Σίγουρα θα επηρεάσει την ε, δραστηριότητα των αλλιέων στις παράκτητες περιοχές. Ο κύριος Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι έχω πολλούς φίλους αλληλείς και υπάρχει και ένας από το Πόρετς που είναι παιδικός φίλος μου και πάντα έλεγε ότι οι αλληλείς έχουν αμφιβολίες και δεν εμπιστεύονται τους νομοθέτες. Θα ήθελα και εγώ να μπω στη θέση του και να εκφράσω αμφιβολίες, γιατί δεν ξέρω πώς θα τελειώσουν όλα αυτά. Θα ήθελα να πιστέψω ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης σημαίνει διατηρήσιμη αλληλεία και αλλιεύματα, αλλά έχω αμφιβολίες ότι θα συμβεί αυτό. Πάντως θέλω να μιλήσω για την ανάγκη να κατησχύσει η αρχή ευελιξίας και η μεταβατική ε, περίοδος. Αυτά τα δύο μπορεί να διευκολύνουν τους αλληλείς να νιώθουν καλύτερα κάποια χρόνια αφού τεθεί σε ισχύ αυτή η οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ένα λεπτό. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι απορρίψεις ε, ψαριών όταν δεν μπορούν να επιβιώσουν δεν είναι βιώσιμοι και δημιουργεί προβλήματα. Πολλοί είναι οι λόγοι, έλλειψη εμπορικής αξίας κάποιων αλλιευμάτων, αλλά υπάρχουν και ανεπαρκή μέτρα διαχείρισης. Θα πρέπει να δούμε την ποικιλία καταστάσεων που μπορεί να προκύψει στον κλάδο της αλληλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για μικρής κλίμακας αλληλεία ή αλληλεία πολλών ειδών, αυτό είναι ένα θέμα. Έχουμε και την βιομηχανική κλίμακα όμως της Ελίας, κυρίως στο Βορρά. Τα προβλήματα που προκύπτουν πρέπει να απαντηθούν. Η Επιτροπή Αλίας έστειλε την προσωπία στις Αζόρες για να παρακολουθήσει το θέμα διατήρησης ε, των σκαφών, βιωσιμότητα κλπ. Μετά τις Αζόρες ε, καταγράψαμε κάποιες τροπολογίες για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Τα οι περισσότερες δεν θεωρήθησαν ε, ε, αποτελεσματικές και απορρίφθησαν. Επόμενος. Ε, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Πρόκειται για έναν κανονισμό ο οποίος ακολουθεί οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι τόσο σαφή τα πράγματα όσο προσπαθεί να μας αποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλές φορές δίνεται εντύπωση ότι αυτοί οι κανόνες ε, είναι μάλλον ε, μακριά από την πραγματικότητα και αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό πραγματικά θα μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε όλες αυτές τις δράσεις. Υπάρχει περίπτωση οι κανόνες αυτοί να προκαλέσουν περισσότερη ζημιά από ότι όφελος. Αναφερθήκαμε στην εποπτεία, στη συνεργασία με τους παρατηρητές και το καθεξής, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και με τους αλληλείς. Θα πρέπει να γίνουν ε, ε έρευνες, να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία και να φροντίσουμε η αλληλεία πραγματικά να είναι βιώσιμη. Και αυτό φυσικά χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος ε, έχει το λόγο. Ή δυνατόν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πολλοί από εσάς αντιμετωπίσατε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Όλοι έχουμε κοινό συμφέρον, το οποίο είναι να ενισχύσουμε και να κάνουμε βιώσιμη την αλληλεία. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε το σημαντικό αυτό τομέα κλάδο της ελίας. Όπως ε, είπαμε, η μετάβαση είναι από την απόρριψη στην ε, εκφόρτωση αλλιευμάτων. Απότερος στόχος είναι να μειώσουμε μέχρι εξαλείψεως των αλλιευμάτων, όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή, ένας τρόπος είναι να ε, έχουμε πιο επιλεκτικό εξοπλισμό και βέβαια αυτή η υποχρέωση εκφόρτωσης προάγει αυτή την ιδέα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι όταν προστατεύουμε τον κλάδο αυτό το κάνουμε προς το βέλτιστο συμφέρον μας και προς το συμφέρον της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των ίδιων των αλλιέων. Κάποιοι μιλήσατε για την ανάγκη ευελιξίας, η οποία ε, υπάρχει στις διατάξεις de και θα προσαρμοστούν για να λάβουν υπόψη και τα τις απορρίψεις. Πολύ μιλήσατε για το όμνιμπους, το πολυνομοσχέδιο που είναι προσωρινό. Η μεταρρύθμιση των τεχνικών ε, μέτρων ε, ε, θα ακολουθήσουν και η αναθεώρηση των υποχρεώσεων θα ακολουθήσουν. Δεν θα αφήσουμε μόνους τους αλληλείς. Υπάρχει υποστήριξη ε, για τους αλληλείς όπως δηλαδή η βοήθεια να αλλάξουν τον εξοπλισμό, να αντιμετωπίσουν τα λιεύματα και στην ξηρά και επί των σκαφών. Ε, κύριος ε, Καντέκ μίλησε για το νομικό θέμα που υπάρχει μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν πρέπει να επανέλθω. Περιορίζομαι σε ένα σχόλιο. Αυτό ήταν ένα θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο. Είμαι ευτυχής όμως διότι το Συμβούλιο ενέκρινε την πλήρη ε, συνολική προσέγγιση. Δεν δημιουργήσε πρόβλημα νομικής βάσης και η Κομισιόν βεβαίως ε, ε, τηρεί τα αποτελέσματα της διοργανικής Task Force. Ανέφερα όλους τους παράγοντες που πρέπει να αναλάβουν με σοβαρότητα την, τις ευθύνες τους για να υπάρχει καλή συνεργασία. Ε, οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει σε τοπικό επίπεδο σίγουρα ε, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα ο εισηγητής, ε, ο κύριος Αλέν Καντέκ, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Merci, Madame la Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ για την ποιότητα της συζήτησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στην εκπόνηση της εισήγησης, τους σκιώδεις εισήγητες, την Γραμματεία, ε, την Επιτροπή, την Λετωνική Προεδρία. Χωρίς όλους αυτούς δεν θα ήταν εφικτή αυτή η εισήγηση. Ευχαριστώ επίσης τους βοηθούς μου Εμιλή και Βενσό θα χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη όλων αν θέλουμε αυτή η εκφόρτωση ε, να λάβει χώρα από αυτό εξαρτάται η αξιοπιστία μας. Ελπίζω η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής των Κρατών Μελών του Κοινοβουλίου, των επαγγελματιών, των επιστημόνων θα επιτρέψει ε, μια ε, καλή εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης ε, προς όφελος του πόρου αυτού και των αλλιέων, διότι νομίζω ότι αυτό θα είναι δύσκολο, όπως το είπα στην αρχή, και ότι η επιλεκτικότητα είναι η πραγματική απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καντέκ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο.